το τέλος των συζητήσεών μας. Περνάμε τώρα στην κατάσταση στο Νεπάλ μετά το σεισμό. Και το λέω έχει ο κύριος Καστάλντο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ανθρωπιστικό δράμα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός στο Νεπάλ είναι τρομερό. 8.800 νεκροί και 22.300 τραυματίες, 814.000 άτομα έχουν χάσει το σπίτι τους και εκατομμύρια χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια και πολύ περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια. Τι συμβαίνει λοιπόν στο Νεπάλ, θα αρχίσει η περίοδος των μουσώνων τις επόμενες εβδομάδες και Δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο με, με, την, με τον ανεφοδιασμό όλων αυτών των, ε, των, των χωριών που χρειάζονται τη βοήθεια, αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε ε, τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει με, τη, με, με την σπορά. Ε, θα, υπάρχει όλη η φετινή εισοδιά. Επομένω θα πρέπει να ε, εκταμιεύσουμε ό,τι μπορεί. Υπάρχει διάθεσή μας. Διακόπτει τον κύριο Καστάλτο η πρόεδρο, Να μιλάτε λιγότερο γρήγορα παρακαλώ, λέει η πρόεδρο. Καλά, καλά, λέει ο κύριος Καστάλτο. Οπότε θα πρέπει ακριβώς όπως έλεγα να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι πόροι υπάρχουν διαθεσή μας να χρησιμοποιηθούν και με διαφάνεια, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επίση οι πιο αδυνατοί να προστατευτούν τα δικαιώματά τους, οι ασθενείς, οι γυναίκες και οι ανήλικοι. Ο κύριος Δεμές για λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχει περάσει 1,5 μήνα από τον καταστροφικό σεισμό και τώρα έχουμε μια καλύτερη εικόνα του πώ χορηγείται βοήθεια στο Νεπάλ και τη δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός. Είναι απίστευτο ότι η αρχή του Νεπάλ εξακολουθεί να εφαρμόζει γραφειοκρατικές διαδικασίες και επιβάλλει δασμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι χρειάζεται να ε, περπατήσουν δεκάδες χιλιόμετρα για να λάβουν βοήθεια. Και η Ντάλιτ που είναι ε, στο κατώτερο σημείο του καθεστώτος καστών που υπάρχει εκεί αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα. Εάν δεν είναι πιο αποτελεσματική η διεθνής βοήθεια, η ανοικοδόμηση της χώρας θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Το ίδιο το κράτος πρέπει να ανοικοδομηθεί νέες δομές με αποτελεσματική ε, διακυβέρνηση σε τοπικό και γενικό επίπεδο και εκδημοκρατισμό τη εκπαίδευση και τη υγεία. Μόνο έτσι θα μπορέσει να έχει θετικέ επιπτώσει αυτή η καταστροφή με τη βοήθεια τη Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Κανέτσνα. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Οποιαδήποτε φυσική καταστροφή είναι τα τραγωδία που οδηγεί σε απώλεια ζώων και καταστροφή της περιοχής. Ε, όταν ε, συμβαίνουν αυτές τις φυσικές ε, καταστροφές σε σημεία όπως η ΑΕΤ και το Νεπάλ μένουμε αναδύ και ανίκανοι να αντιδράσουμε. Δεν υπάρχει αστικοποίηση, ούτως ή άλλως πλήττεται από τη φτώχεια η αλλως πληττει απο τη φτωχεια η περιοχη και πάνω από 8 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται πλέον ανθρωπιστική βοήθεια. Σίγουρα υπάρχει παροχή τοπικής βοήθειας, όμως πρόκειται για απελπισμένους ανθρώπους που χρειάζονται την βοήθειά μας, κυρίως σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, θα πρέπει να ε, παρασχεθούν παραδείγματο χάρη ιατρικέ ε, σκηνέ, ε, διότι δεν υπάρχει πλέον υποδομή ιατρική περίθαλψη. Ε, είναι καθήκον της διεθνούς κοινότητας να φροντίσει για την επανένωση των παιδιών με τι οικογένειε του, παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στα παιδιά, διότι βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση ε, υπά, ο λοιμός ε, αλλά και δυστυχώς η εμπορία παιδιών είναι καθημερινά φαινόματα βάσει ε, των ε, ε, ομάδων που δρούν επί τόπου. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να φροντίσει ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να μπορέσει με συστηματικό τρόπο να φτάσει σε αυτούς που τη χρειάζονται, καταργώντας τους φραγμούς που προβάλλει ορισμένες φορές η αστυνομία επί τόπου. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί ε, το, το, το βασανιστήριο αυτό για, τους, για τον ε, εγχώριο πληθυσμό. Θα πρέπει ε, να δράσουμε αμέσα διότι υπάρχουν, υπάρχει ο κίνδυνος των μετασυσμικών δονήσεων. Σας ευχαριστούμε κύριο Σμάνη ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις αρχές Απριλίου μια μέλη της αντιπροσωπής για την Νοτιοανατολική Ασία πήγαμε στο Νεπάλ και θέλαμε να θαρρύνουμε τους ε, προέδρους των ε, σημαντικών κομμάτων να αποφασίσουν για ένα ψήφισμα για την αλλαγή του κλίματος και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν επιτύχει σημαντικές ε, πρόοδους. Και επισκεφτήκαμε και ένα πρόγραμμα της Ένωσης, ένα νοσοκομείο. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι δύο αργότερα θα πέθαιναν 9.000 άτομα. Από αυτόν τον τρομερό σεισμό εκατοντάδες χιλιάδες έχασαν το βιό τους και τα σπίτια τους και τρομερά πολιτιστικά μνημεία στην Κατμαντού και στον Πακταπούρ που τα είχαμε επισκεφτεί δεν υπάρχουν πλέον. Το κύμα τη αλληλεγγύη είναι εντυπωσιακό. Χιλιάδε εθελοντέ βοηθούν και οι παραδοσει ε, τροφίμων και φαρμάκων και οικονομική βοήθεια έχουν όλα ανέλθει για παράδειγμα από τη Γερμανία 60 εκατομμύρια σε μερικέ εβδομάδε, όμω σε τέτοιε περιπτώσει των μηνιών οι τοπικές αρχές και το σύστημα υγείας πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά ώστε το συναρπαστικό Νεπάλ με το οποίο είμαι συνδεδεμένος εδώ και δεκαετίες να μην μείνει μόνο του για να αντιμετωπίσει. Να είμαστε! Ο κύριος ε, Λαμπέρτ για ένα... Η κυρία Λάμπερτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, Προεδρεύω στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, στην οποία αναφέρθηκε μόλι ο κ. Μαν που πήγε στο Νεπάλ ε, δύο εβδομάδε πριν ε, χτυπήσει ο σεισμό. Ξέρουμε ότι εφαρμόζονταν προγράμματα για τη μετώπιση φυσική καταστροφή, αλλά όχι σε ολόκληρη την επικράτεια. Ξέρουμε όμω ότι χάρη σε αυτέ τι προετοιμασίε σώθηκαν ζωέ. Παρ' όλα αυτά, να εκφράζουμε την συμπόνια και την αλληλεγγύη και τα συλληπιτήριά μα προ αυτού που έξαν του αγαπημένου του και προ το σύνολο τη χώρα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα υλικοτεχνική επιμελητία ε, για την ε, παροχή ανθρωπιστική βοήθεια ε, λόγω γεωγραφικών λόγων και καθυστερήσεων ω προ την ανάπτυξη τη χώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη συμφωνία, διακομματική συμφωνία για το νέο σύνταγμα καθώ και την ανακήρυξη τη νέα κυβέρνηση, η δράση τη οποία θα είναι απαραίτητη για την ανόρθωση τη χώρα. Το ΑΕΠ τη χώρα δεν θα μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά διότι ο τουρισμός είναι το βασικότερο, η βασικότερη πηγή εισοδήματος και ε, ε, το κόστος ε, των σημείων αντιστοιχεί σε το 50% του ΑΕΠ. Ευχαριστούμε. Διακόπτη η Πρόεδρος, η κυρία Σαράνσοβα. Ένα λεπτό. Τον σε διαρκεί. Κατάσταση κατεπηγούσης ανάγκης, οπότε θα πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να θεωρηθεί ότι χρειάζεται και αυτή η συνέχεια να βοηθήσουμε την συγκρότηση αυτή τη πανέμορφη χώρα που είχα την τιμή μία φορά να επισκεφθώ. Βέβαια, στο επίκεντρο των προσπαθειών θα πρέπει να βρίσκεται σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυστυχώ έχουμε πάρα πολλέ καταγγελίε ότι οι πιο κοινωνικέ ομάδε τίθενται ε, διακρίσει ε, δυσμενεί επί τη βάση του φίλου του ή τη ε, θρησκεία του. Οπότε θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, όλο και τον ε, πληθυσμό και θα πρέπει η βασική βοήθεια να πάει σε όλους ε, ανεξαρτήτως από την προέλευσή τους. επίσης αυτή η τραγωδία χτύπησε και τα παιδιά. Έχουμε πάνω από 7.000 σχολεία τα οποία αγκρεμίστηκαν οπότε θα πρέπει και αυτά να ξαναχτιστούν σαν προτεραιότητα. να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι καθήκον μας και να ξαναγυρίσει στην ομαλότητα η χώρα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ο κύριος Καν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και εγώ πήγα στο Νεπάλ δύο εβδομάδες ε, πριν από την τραγωδία και βλέποντας τις εικόνες καταστροφής των περιοχών που είχαμε επισκεφθεί, μουράγισε την καρδιά 2,8 εκατομμύρια ε, ζητούν, ε, χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και ένα εκατομμύριο είναι σε δυσπρόσιτες περιοχές. πριν προκληθούν και άλλες ζημιές, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές. επίσης, για οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια παρέχεται, πρέπει να εξασφαλιστεί ισότιμη ισότιμη πρόσβαση και κυρίως ισότιμη κατανομή προς όλους. Ε, όπως τόνισε ο ΙΕ, χρειαζόμαστε όμως αύξηση τη ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό που χρειάζεται τον πάλι είναι πακέτο βοήθειας ε, για την ε, ανασυγκρότηση της χώρας, ε, καθώς και ένα εθνικό πρόγραμμα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστραφών. Η περιοχή του Κατμαντού φυσικά θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο σε αυτές τις προϊούσες προσπάθειες για να επιτευχθεί η ειρήνη και η ευημερία και ελπίζουμε να ενωθούν Όλε όλες ε, οι δυνάμεις από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, διότι χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ ε, την πολιτική συνένεση. Σας ευχαριστούμε τώρα από πλευρά των πολιτικών ομάδων. Κυρία Τούνε, δεν σας έβλεπα, δυσκολεύτηκα να σας βρω με στην αίθουσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τραγικές ε, εικόνες από τον ΕΠΑΛ Είδε ολόκληρος ο κόσμος ε, πριν από λίγες εβδομάδες ε, μετά το σεισμό, όμως ε, το πρόβλημα είναι και όσοι έχουν πάει στο Νεπάλ το ξέρουν, ξέρουν ότι πέρα από την απαράμιλη ομορφιά του τοπίου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που πλήττουν τον εγχώριο πληθυσμό και ε, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ε, όπως ε, αυτός ο σεισμός οξύνονται τα στάμενα προβλήματα κυρίως αυτών που ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές. Χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως καλύτερες συνθήκες, πόσιμο νερό, πρόσβαση σε κάποιες περιοχές, πέρα από την αλληλεγγύη θα πρέπει να παραμείνουμε στο πλευρό του Νεπάλ με διαρκή δράση, με παροχή απτής ε, βοήθειας. Διακόπτη, Πρόεδρος. Ε, ε, υπερβήκατε το χρόνο αγόρευσή σας, κυρία μου. Η κυρία Τζιλ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μακροχρόνια σχέση με τον Νεπάλ. Έχω εργαστεί με το κίνημα υπέρ της δημοκρατίας πριν από τις ε, πρώτες ε, παγκόσμι... ε, δημοκρατικές εκλογές στην ιστορία της χώρας. Γι' αυτό θα βάζω ιδιαίτερα το λαό του Νεπάλ και την αποτελεσματικότητά του και την αποφασιστικότητά τους να ξαναχτίσουν τη χώρα τους μετά τον καταστροφικό πρόσφατο σεισμό. Μία από τις κύριες ανησυχίες μου τώρα είναι τα παιδιά. Υπάρχουν 1,7 εκατομμύρια ευάλωτα παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους και πολλά έχουν μετατοπιστεί εσωτερικά. Και γι' αυτό τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα υπ' αυτέ τι συνθήκε. Ότι μπορεί να τα πάρουν ε, ενήλικε που δεν έχουν καμία συγγενική σχέση ή μπορεί να απαχθούν. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν διαδικασίε επιτόπου για να το σταματήσουν αυτό. Και επίση να αναγνωρίσουμε ότι έχουν καταστραφεί πολλά σχολεία. Πρέπει λοιπόν να ενωθούμε και να δώσουμε προτεραιότητα στην ε, ανοικοδόμησή του, ούτω ώστε να γυρίσουν στο σχολείο. Να μην καταστραφεί το μέλλον του. Πρόεδρε, η περίοδος των μουσώνων ξεκινάει και αυτό θα επηρεάσει τις προσπάθειες ανακούφισης. Ευχαριστώ κυρία μου, λέει η Πρόεδρος. Και κόβει το μικρόφωνο. Ο κύριος Κάρσκι από πλευράς των συντηρητικών. Ευχαριστώ πολύ. πάνω από 8.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ε, εκατοντάδες χιλιάδες έχασαν τα σπίτια τους, πολύ περισσότεροι είναι πρόσφυγες. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της τραγωδίας. Αναφέραμε τις προσπάθειες που κάναμε στέλνοντας διάφορους εμπειρογνώμονες, ε, ιατρικό προσωπικό από διάφορες χώρες της Ένωσης. Από την αρχή δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε πολλή βοήθεια. Στείλαμε 40 εκατομμύρια για την άμεση αντιμετώπιση. Και τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε μια συζήτηση και για την ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά και για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ελευθερία. Πρέπει να πούμε ότι οι αρχέ του Νεπάλ πρέπει να εφαρμόσουν πολιτική ε, ευκολότερη ε, πρόσβαση τη ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί την επιβαρύνουν με δασμού και επιπλέον δεν αποστέλλεται εκεί που πρέπει σε όλου. Για παράδειγμα, στι γυναίκε Ντάλιτ Αυτές έχουν θυγεί ιδιαίτερα γιατί δεν πάει σχεδόν τίποτα σε αυτές. Αυτές οι διακρίσεις πρέπει να σταματήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει συνέστηση του τι συμβαίνει. Ευχαριστώ για την άλλη, ο κύριος Γιάκοβτσης, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη η τραγωδία της 25ης ε, Απριλίου, αλλά ο και ο του 5 Μαΐου, οπότε είχαμε ένα εκατομμύριο 1,7 εκατομμύρια παιδιά τα οποία δεν έχουν τον ένα ή και τους δύο ε, γονείς τους. 1,4 ε, ε, εκατομμύρια άτομα έχουν και βοήθειας. Προχωρεί η βοήθεια σύμφωνα με τις, τους υπολογισμούς, μιλούμε για 10 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί ε, το, το πρόβλημα σε σχέση με τα τρόφιμα που θα συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον. Οπότε έτσι θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να δώσει χρήματα και ανθρωπιστική βοήθεια. Ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος να αποκαταστήσει τις ζημίες που έχουν γίνει και επίσης θα πρέπει να προστατεύσουμε και τα μνημεία πολιτιστικής οικονομίας. Ένα λεπτό, η κυρία Λόπες. Όλα αυτά τα οποία αφορούν ε, ανθρώπους και στο Νεπάλ και στο Μίλη στην Παραγουάη δεν μπορεί παρά αυτά να μας αγγίζουν. Δεν μπορεί να τα θεωρούμε ξένα γιατί από ό,τι φαίνεται ο κόσμος γίνεται ένα εχθρικό περιβάλλον και έχουμε αυτές τις ε, θεομηνίες που είναι τόσο συχνές και ε, αναπόφευκτες φαίνεται. Όμως δεν είναι έτσι το Νεπάλ έχει πέσει θύμα της παγκοσμιοποίησης που προχωρεί, το που προωθεί και η Ευρώπη. Έχουμε ένα σωρό μετανάστες εκεί. Ε, οι, ίδιοι οι Νεπαλέζοι έρχονται στην Ευρώπη σαν, σαν ε, πρόσφυγες και ζουν σε τρομερή κατάσταση. Τους πνίγουν οι συνθήκες που επιβάλλει το διεθνές εμπόριο και έτσι δεν είναι δυνατόν να πιάσει τόπο η αναπτυξιακή πολιτική. Είναι κάτι σαν φαύλο κύκλος. Εμεί έχουμε υποχρεώσει αλληλεγγύη, αλλά δεν ε, το κάνουμε αυτό. Έχουμε από τον ΟΗΕ μόνο 300 εκατομμύρια, τα οποία όμω δεν έχουν ακόμα εκταμιευθεί από τον ΟΗΕ. Και το αρχίζει το ΚΑΤΣΔΙ. Έχουν 7 συναδελφιστές στο λόγο. Α, μισό λεπτό κύριε Κέλλη, έχετε εσεί το λόγο. Συμπαθάτε με, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, αναμφίβολα. Είναι ιδιαίτερα λυπηρή η κατάσταση. Είναι λυπηρές συνθήκες υπό τις οποίες ζουν ακόμη οι άνθρωποι στο Νεπάλ. 9.000 νεκροί, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς σπίτι, τα σχολεία καταστραμμένα. Πρέπει λοιπόν να τους βοηθήσουμε. Και η Επιτροπή έχει στείλει ε, βοήθεια και οι Ηνωμένε Πολιτείε 10 εκατομμύρια και η Βρετανία έχει στείλει 6 εκατομμύρια λίρε. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν το ερώτημα. Η βοήθεια αυτή φτάνει εκεί που τη χρειάζονται περισσότερο. Ιδιαίτερα στην κοινότητα των Ντάλιτ. Ε, αυτή που είναι στο χαμηλότερο σκαλί της ιεραρχίας ε, των καστών. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι αυτή η βοήθεια φτάνει στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Άλλο θέμα Μήπω έχουμε πολλές, υπερβολικά πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις επιτόπου. 16 έχω ακούσει. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι λιγότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό θα βοηθούσε. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει η διαδικασία ε, προσέλκυση προσοχή του Προέδρου. Ο κύριο Σόγκορ, πρώτο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, οι Νεπαλέζοι έζησαν ε, πάρα πολύ δύσκολες ε, στιγμές το περασμένο μήνα με αυτή την τραγωδία του σεισμού και θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Υπάρχουν χιλιάδες Θηβετιανοί πρόσφυγες που ζουν στο Νεπάλ και δεν έχουν ως επιτοπλίστων την υπηκότητα και άρα δεν υπάρχουν στα μάτια του κράτους. Οι Θιβετιανοί στο Νεπάλ δεν έχουν εγγυημένα τα βασικά τους δικαιώματα διότι στο Σύνταγμα του Νεπάλ εφαρμόζονται τα δικαιώματα μόνο για τους πολίτες. Επίσης δεν είναι και μέρος στη Σύμβαση για την προστασία του καθεστώτος του πρόσφυγα. Βλέπουμε ότι σε τέτοιες στιγμές ε, πόσο ξεκάθαρο είναι ότι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού εκτίθενται στα μεγαλύτερα προβλήματα και θα πρέπει λοιπόν οι αρχές του Νεπάλ να ε, κάνουν τα απαραίτητα ώστε σε περίπτωση κρίσης όπως σε συγκεκριμένη περίπτωση να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα όλων ακόμη και αυτών που δεν έχουν την υπηκότητα. Ευχαριστούμε. Ε, θα καλούμε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες ανασυγκρότησης ε, στο Νεπάλ και να αυξήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στη χώρα. Θα ήθελα να εκφράσω τα ε, συλληπιτήριά μου προς τις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη μου προς τους Νεπαλέσους μετά τον καταστροφικό σεισμό και τους μετασυσμούς στη χώρα. Να ευχαριστήσω επίσης το κράτος του Νεπάλ καθώς και την διεθνή κοινότητα για τις προσπάθειες που έκαναν για την ανασυγκρότηση. Αληθεύει όμως ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για τις ε, επιχειρήσεις ε, έρευνας και διάσωσης ε, και να σώσουμε αυτούς που βρίσκονται σε δυσπρόσθετες περιοχές, να υπάρχει ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων στην ανθρωπιστική βοήθεια και να λάβουμε μέτρα για μεγαλύτερη εντοχή της χώρας και άμβληνση των επιπτώσεων τέτοιων κρίσεων. επίση, στο τομέα τη Δημοκρατία μέσω τη αναπτυξιακής βοήθεια μπορούμε ε, να επιτύχουμε πολύ περισσότερο. Κύριε Μαριέ. Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζω το δράμα των σεισμόπληκτων, τι αγωνίε του και τι ανάγκε του, καθώ η πατρίδα μου η Ελλάδα έχει πληγεί συχνά από τον εγκέλαδο. Στο Νεπάλ οι σεισμοί οδήγησαν σε 9.000 νεκρού και σε χιλιάδε τραυματίε. Ταυτόχρονα 2,8 εκατομμύρια συνάνθρωποι μα αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική κρίση χρειάζεται λοιπόν αυξημένη διεθνής βοήθεια και αλληλεγγύη στο νεπάλ. πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό με σκηνές σε πρώτη φάση και ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης στη συνέχεια. η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι απαραίτητη όπως επίσης και η επιστημιστική βοήθεια. η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει παντού σε όλες τις δυσπρόσιτες περιοχές σε όλους τους σεισμόπληκτους εκατομμύρια παιδιά στο νεπάλ έχουν χάσει τους γονείς τους και πρέπει να διαμορφωθεί ένα δίκτυο προστασίας των παιδιών για να μην απαχθούν από τους δουλέμπορους. κυρία πρόεδρε το νεπάλ εκπέμπει σως και η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα με ακόμη μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα τη συζήτηση. Φυσικά και πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα. Αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την δίκαιη κατανομή της βοήθειας. Να μην υπάρχουν δυσμενεί διακρίσεις και κάποιοι να μείνουν χωρίς αυτή τη βοήθεια. Θα πρέπει να πιάσει τόπο η προσπάθεια βοηθεια όπω και άλλοι συναδελφικοί συγκλονιστή, αυτά που διαβάζω στον τύπο. Επίση, έχουμε και τι μαρτυρίε των Τσέχων εθελοντών που έχουν εσπεύσει εκεί. Υπάρχουν κάποιε κοινωνικέ ομάδε που δεν παίρνουν καθόλου βοήθεια. Πρόκειται για κάποια φτωχά παιδιά, κάποιε γυναίκε, κάποιε μειονότητε και γι' αυτό χαίρομαι που ε, απευθύνουμε έκκληση στην κυρία στο κείμενό μα να ξεκινήσει επαφέ με την κυβέρνηση τη χώρα. Να εξασφαλίσει τη δίκη μοιρασιά τη βοήθειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλιώ θα γίνει η βοήθεια παιχνιδάκι στα χέρια των ισχυρών της χώρας. Πώς ε, σας εύχομαι χρόνια την γενέθλιά σα, Πρόκειται για μια τραγωδία στη χώρα που έχει ελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου. Έχει πεθάνει πολλοί κόσμος, κάποιοι έχουν μείνει ε, άστεγοι, ε, λείπουν φάρμακα και είδη διατροφής. Άρα θα πρέπει όλους αυτούς να τους ε, βοηθήσουμε. Έχουν πάει πολλοί εθελοντές και από τη δική μου χώρα εκεί, οπότε θα πρέπει η Ένωση και το Κοινοβούλιο να δείξει αλληλεγγύη. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Οπότε θα πρέπει επίσης να δούμε με τι άλλους παραπάνω τρόπους θα βοηθήσουν τον κόσμο εκεί. Όλους αυτούς οι οποίοι πεθαίνουν ε, έξω στο δρόμο, δεν έχουν ε, σπίτι. Παρακαλώ πιο αργά, λέει πρώτα στην ομιλήτρια. Έλεγα, κύριε Πρόεδρε, ότι το 1997 στη χώρα μου είχαμε ένα σημαντικό σεισμό. Ο σεισμός αυτός άφησε πάρα πολλούς άστεγους. Οπότε δεν μπορούμε παρά να δείξουμε αλληλεγγύη προς το Νεπάλ. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να δείξει αλληλεγγύη. Μιλήσατε πάρα πολύ γρήγορα, λέει ο Πρόεδρος. Έχει το λόγο τώρα η κυρία Σουίκα για ένα λεπτό. Ε, Μα έχει ε, καταθλίψει αυτό που μαθαίνουμε για αυτά που συμβαίνουν ενάμιση μήνα μετά την ανθρωπιστική τραγωδία, την καταστροφή. Πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε επαρκεί πόρου και πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, σωστή και διαφανή χρήση αυτών των πόρων. Η κυβέρνηση του Νεπάλ ζητά ακόμη ανθρωπιστική βοήθεια. Ξέρουμε ότι και πριν από την τραγωδία ούτω ή άλλως η χώρα ήταν ε, φτωχή, ε, υπανάπτυκτη και 50% του ΑΕΠ της ε, προέρχονταν από τον τουρισμό, ο οποίος τώρα θα μειωθεί. Γι' αυτό πρέπει να χορηγήσουμε βοήθεια στα εκατομμύρια που την χρειάζονται. Και το ψήφισμα αυτό είναι η δυνατότητα να καλέσουμε τα κράτη-μέλη της Ένωσης να βοηθήσουν. Πρέπει να επιδείξουμε έμπρακτη αλληλεγγύη, να μην νομίζουμε ότι τον Νεπάλ είναι πολύ μακριά. Μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Και τέλος η κυρία Ταπάρντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε περίπτωση κρίσης ε, θα πρέπει να συνεργάζονται όλοι και να δείχνουν την αλληλεγγύη τους και να πανεμβαίνουν υπέρ αυτών που χρήζουν βοήθειας. Ε, το ένστικτο βοήθειας ε, προς όσους το χρειάζονται είναι μια βασική αξία του ανθρωπίνου είδους. Χρειάζεται να δείξουμε αλληλεγγύη προς την κοινότητα αυτών των ανθρώπων που πλήττεται από τα ανεξέλεγκτα φυσικά αυτά φαινόμενα. Στις 13 ε, Μαΐου μετά το σεισμό 1,7 παιδιά έχουν μείνει αβοήθητα. Έχει σβήσει το μικρόφωνο Κυρία Καπερδέλη, μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, παρακαλώ να επιβραδύνετε. Ε, χρειάζεται τριπλασιασμό των πόρων τη ανθρωπιστική ε, βοήθειας. Έχει ήδη αυξηθεί, όμως δεν αρκούν αυτά. Πρέπει να συνεργαστούμε ούτω ώστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι να ε, βοηθήσουμε τον λαό του Νεπάλ να δώσει την απαιτούμενη βοήθεια στους πολίτε στο κράτο. Τώρα θα ε, πάρουμε, θα ακούσουμε την κυρία Καλινίτσα Σεβίτσα, εξ ονόματο ε, της κυρίας Μογκερίνης, είπα της εκπροσώπου και αντιπρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδες για τι εξωτερικέ υποθέσει. Ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξ τη ε, της είπα τη εκπροσώπου κυρία Μογκερίνη. Θα ήθελα να καλωσορίσω την υιοθέτηση της, του κατεπήγοντο ψηφίσματος του Κοινοβουλίου για την κατάσταση στο Νεπάλ μετά του καταστροφικού σεισμούς Στι στις 25 Απριλίου και 12 Μαΐου. Υπάρχει μια στενή σχέση φιλίας ε, που ενώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της με τον ΕΠΑΛΗ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της ε, έχουν ήδη εκφράσει την ε, συμπόνια και αλληλεγγύη τους για τις ε, απώλειες ανθρώπινων ζώων ε, και βλαβών ε, καταστροφών των σπιτιών της υποδομής και τόπων εθνικής κληρονομιάς στον Ιπάλ. Δεν έχουμε λόγια για να περιγράψουμε το, την κλίμακα αυτής της τραγωδίας. Ταχύτατα αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της και έδειξε αυτή η αλληλεγγύη προς το λαό του Νεπάλ. Αμέσως μετά το σεισμό και μετά από την έκκληση που μας κυβέρνηση του Νεπάλ σαφέστατα Καταδείξαμε την αλληλεγγύη μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρίσχε 3 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για να υποστηρίξει κυρίως ε, κατεπίγουσες ε, την κατασκευή ε, καταβλισμών, την παροχή ιατρικής περίθαλψης και την υλικοτεχνική επιμελητία και συντονισμό. Επίσης, διπλασιάσαμε αυτό το ποσό στα 6 εκατομμύρια μετά την επιτόπου επίσκεψη του Επιτρόπου Αρμοδίου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια του Χρήστου Στυλιανίδη, ο μαζί με τη Βαλερία Μος, την Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ, αρμόδια για τον συντονισμό της ε, άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, μετέβησαν στον ΑΠΑΛ για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Ε, και επίσης ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε άμεσα, ότως ώστε τάχιστα να παρασχεθεί και υλικό για την ανακούφιση, καθώς και αρρωγή εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίση υπήρξε και μέσω των προξενείων υποστήριξη προς τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νεπάλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιτάχυνε την εκταμείευση 16,6 εκατομμυρίων από τα αναπτυξιακά ταμεία. Αυτή η πρόερη ε, εκταμείευση συγγνώμη, επιτρέπει στις αρχές του Νεπάλ να ανταποκριθούν στις πλέον κατεπίγουσες ανάγκες. αξιότιμοι βουλευτές. Επίσης, εξετάζουμε το ενδεχόμενο χρήση άλλων ε, ε, εργαλείων που έχουμε για να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση της σταθερότητας και της ειρήνης, ε, παρέχοντας έτσι τα απαιτούμενα εφόδια στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές που είναι και δυσπρόσιτες. Έγιναν δυσπρόσιτες μετά το σεισμό. Ε, χρειαζόμαστε επίσης επιρρόσθετη υποστήριξη για την χώρη Φίτηση σε σχολεία έχουν καταστραφεί από το σεισμό. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για την τρέχουσα κατάσταση βάσει του μνημονίου συνεννόησης. Ε, ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι, με συγχωρείτε. Συνάδελφοι, καταλαβαίνω γιατί μπαίνετε τώρα αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Σας παρακαλώ όμως ε, να ε, ε, το κάνετε ίσχα και χωρίς θόρυβο, διότι από για την ομιλήτρια. Αξιότιμοι βουλευτές. Μιλάμε για τον σεισμό στο Νεπάλ και ε, εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ε, ε, μιλάμε για τα, τους τελωνιακούς δασμούς, υπάρχει ένα μνημόνιο συνεννόησης που πριν από πολλά χρόνια υπεγράφει με τον Νεπάλ και ατέλεια εισέρχονται έτσι εφόδια ανθρωπιστικής βοήθειας ε, στο Νεπάλ. Λίγες ημέρες ε, μετά το σεισμό η κυβέρνηση του Νεπάλ ε, υιοθέτησε αυτή την προσέγγιση μετά και την επίσκεψη του Επιτρόπου Στυλιανίδη που δρομολόγησε όλες αυτές τις διαδικασίες. Παραμένουν, ε, παραμένει λοιπόν ε, η δασμολογική ατέλεια για, για την ανθρωπιστική βοήθεια από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ε, συλλέγονται συστηματικά πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας ε, και ε, αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν ως τεκμηρία ώστε να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τυχόν προβλήματα από πλευρά του ΙΕ. αν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ανακύψουν άλλα κολλήματα θα συνεργαστούμε στενότερα με την κυβέρνηση του Νεπάλ μετά τις επαφές που κάναμε στην πρώτη ανταπόκριση μετά το σεισμό. Τώρα ε, ε, ιδιαίτερα ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει και στην αξιολόγηση της κατάστασης μετά την καταστροφή στα μέσα Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί από ό,τι προβλέπεται και θα αποτελέσει και τη βάση της ε, στρατηγικής αποκατάστασης. Επίσης θα συμβάλλουμε στην συνδιάσκεψη δωρητών που θα γίνει στο Κατμαντού στις 25 Ιουνίου. Σας ξανδιακόπτω, ζητώ συγγνώμη. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ομιλήτρια και μην θορυβείτε. Καθίστε παρακαλώ. Αξιότιμοι βουλευτές, ε, τον Νεπάλ επίσης χρειάζεται πολιτική σταθερότητα ε, για να μπορέσει να προωθήσει την ε, οικονομική μεγέθυνση ε, του και την ανασυγκρότηση της χώρας. Το νέο σύνταγμα μπορεί να υιοθετηθεί άμεσα ως ένα βασικό βήμα στην ειρηνευτική διαδικασία. Στη συνέχεια θα, ακολουθήσουν, θα ακολουθήσει η συγκρότηση πιο αποκεντρωμένων θεσμών με μεγαλύτερη λογοδοσία και έτσι θα αποκατασταθεί και αξιοπιστία σε τοπικό επίπεδο επίπεδο των ΕΜΑΛ επίση ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσει βασικέ προκλήσει σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα να ε, εξασφαλιστεί η ισότιμη απονομή δικαιοσύνη σε όλους τους σεισμόπληκτους ε, ανεξάρτητα με το αν έχουμε την υπηκότητα ή όχι. Ε, μη διακριτικές μεταχειρήσεις ε, ε, λόγω εθνοτικής προέλευσης, προστασία των ανθρωπίνων, των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτά είναι βασικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει τον ΕΠΑΛ, διότι παρατηρείται βία κατά των γυναικών και χρειάζονται καλύτερες κοινωνικές συνθήκες και προστασία, διαφύλαξη των δικαιωμάτων δικαιωμάτων των Έχει αναλάβει μέτρα ε, η κυβέρνηση του Νεπάλ για να βαρεποδίσει το εμπόριο των παιδιών, τα παγωγή και εμπόριο παιδιών. Μετά το σεισμό, παραδείγματο χάρη, παρακολουθεί στενά την κατάσταση η κυβέρνηση του Νεπάλ και ε, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε αυτό, στις πλέον στις πιο σοβαρά στι περιοχέ έχουν σημειωθεί περιστατικά απαγωγών και εμπορία μικρών κοριτσιών. Ήδη σα παρακαλώ μη θορυβείτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορε ανθρωπιστικέ οργανώσει που ασχολούνται με την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών και με το εμπόριο ανθρώπων δραστηριοποιούνται και εμεί έχουμε χρηματοδοτήσει από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωσης προγράμματα για να αντιμετωπίσουμε ε, συγκεκριμένα περιστατικά αλλά και ε, την ε, υποστηρίξουμε τι οργανώσεις των Νταλή που βρίσκονται χαμηλότερα στο σύστημα των καστών καθώ και ε, τους κατοίκους των παραγκοπόλεων αλλά και τις γυναίκες και τα παιδιά γενικότερα. Πέρα από την ε, κατανομή της ανθρωπιστικής ε, βοήθειας προσπαθούμε ταυτόχρονα να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία και να εξασφαλίσουμε η ισότιμη κατανομή της βοήθειας. Είναι ανίποτη η τραγωδία που έπληξε τον ΕΠΑΛ και θα χρειαστεί χρόνος για την πλήρη ανασυγκρότηση της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς εταίροι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον Νεπάλ και το λαό του σε αυτήν την ε, Ηράκλεια προσπάθεια. Σα ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την κατάσταση στον Νεπάλ. Σα ευχαριστώ. Α, από ό,τι φαίνεται ορισμένοι σα άκουσαν κύριε Πρόεδρε. Έχω λάβει 7 προτάσει ψηφίσματος για να κλείσει αυτή η συζήτηση, η οποία μόλι έκλεισε και η ψηφοφορία θα γίνει στο τέλο των συζητήσεων, δηλαδή σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι. Θα αρχίσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ καθίστε. Παρακαλώ καθίστε και βάλτε τις κάρτες σας παρακαλώ στο μηχάνημα. Ευχαριστώ. Έχει γίνει μια δήλωση για προσωπική, μια ένα αίτημα για προσωπική δήλωση. Η κυρία Πυρίνσκι έχει το λόγο. Mr. you have the... Ο κύριος Πυρίνσκι έχει το λόγο. working. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την έκθεση της, ε, του Εποπτικού Συμβουλίου της Εποπτικής Επιτροπής για το Όλαφ, ο κύριος Σαρβράμα, μέλος του Κοινοβουλίου, θύνηκε προς εμένα με τους πιο προσβλητικούς και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Είπε ότι λέω εσκεμμένα ψέματα ότι συνειδητά προσπαθώ να παραπλανήσω το σώμα με τον πιο συκοφαντικό τρόπο. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου εντελώς απαράδεκτο και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων των συναδέλφων από αυτού σε όλες μου τις προσπάθειες. Έχω εκφράσει σαφείς απόψεις, αλλά από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι είμαι σε θέση να καταλάβω, παρουσιάζουν τα γεγονότα όπως τα αντιλαμβάνομαι. Θα συνεχίσω αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού όπου μπορώ να εισέλθω στην ουσία των θεμάτων γιατί ξέρω ότι δεν το επιτρέπει αυτό το άρθρο 164 του κανονισμού αλλά θέλω να είμαι απόλυτα σαφής ότι το είδος της διαδικασίας που θα γίνει στην, που ακολουθείται στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού πρέπει να αναθεωρηθεί και να αναβαθμιστεί σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν γίνει μια σειρά από για δηλώσεις και αντιδράσεις. Οπότε σας παρακαλώ να έχετε υπομονή. Οπότε, κύριε Σαρβάμα, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πυρίνσκι, σας ζητώ συγγνώμη για την ε, ορολογία που χρησιμοποίησα όσον σας αφορά. Τους όρους που χρησιμοποίησα. Ο λόγος ήταν ότι νομίζω ότι γνωρίζω ότι έχετε ε, τη δυνατότητα να γνωρίζετε ότι αυτό που είπατε ότι δεν είχε καμία δυνατότητα η Όλαφ να, να απαντήσει στην ετήσια έκθεσή μας για τη δραστηριότητα της Εποπτικής Επιτροπής. Νομίζω ότι ξέρετε ότι ε, είχε αυτή τη δυνατότητα, αλλά τούτου λεχθέντος ε, σας ζητώ συγγνώμη για τους όρους που χρησιμοποίησα και ελπίζω να τη δεχτείτε τη συγγνώμη. Thank you very much. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Γλέζος, παρακαλώ, για διαδικαστικό. Είχα ζητήσει τον λόγο πριν από την ημερήσια διάταξη. Τους διέφυγε να μου τον δώσουν και μου απάντησαν ότι θα τον δώσουν στο τέλος της ε, ομιλίας. Αυτό δεν έγινε. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω τώρα για αυτό το θέμα που ζήτησα το λόγο πριν από την ημερήσια διάταξη. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Στην σύγκλιτο τη Ρωμαϊκή κάθε πρωί ακουγόταν «Χάνιμπαλ άντε πόρτας» και από μένα κάθε μέρα θα ακούτε κάτω τα χέρια από την Ελλάδα δεν επιτρέπεται να επεμβαίνετε στη χώρα μου που χαράζει ο λαός της το δικό της το δρόμο. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα όσοι υπερασπίζετε τους δανειστές να βοηθάτε τους δανειστές. Η μόνη, Mr. Nuttall, have Η μόνη λύση είναι Oh, Η μόνη λύση είναι να σταματήσει για ένα χρόνο το πάγωμα όλων των υποχρεώσεων της Ελλάδας και ο ελληνικός λαός είναι σε θέση να βρει μόνος του το δρόμο. Ευχαριστώ. Δεν ήταν ακριβώς διαδικαστικό, αλλά σας ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Νάτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μα είδατε τι έγινε χθε το βράδυ εδώ. Αυτό είναι ντροπή. Δυνάμει του 199 ζητήθηκε να διακοπεί η σύνοδος και θα πρέπει να ψηφίσουμε. Εκείνη την ώρα, αντί γι' αυτό, η αντιπρόεδρος ε, ανέλαβε την ευθύνη να κάνει μια διακοπή 30 λεπτών ούτως ώστε και εσείς να έρθετε εδώ να μαζέψετε ένα στον άλλο και να ψηφίζετε. Ε, και για αυτό το λόγο τόσοι θεωρούν ότι εδώ πέρα είμαστε ένα κοινοβούλιο τη πλάκα. Οπότε είτε πάει σοβαρότητα είτε όχι. Ή θα πρέπει κανεί να τηρεί τον κανονισμό είτε όχι. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ό,τι μα βολεύει. Ακριβώ όπω έγινε χθε το βράδυ. Γι' αυτό και θέλουμε ο πρόεδρο Σούλ να διευκρινίσει ότι θα πρέπει ο κανονισμό να ισχύει για κάθε περίπτωση και να μην έχουμε τέτοιε διακρίσει όπω χθε το βράδυ ε, ει βάρο ε, κάποιων οι οποίοι θεωρούνται ευρωσκεπτικιστέ. Well, Mr. Nuttall, um... Όχι, η διακοπή συνεδρίας έγινε γιατί είχε διασυνδευτεί η τάξη σύμφωνα με ε, το άρθρο 22. Φαντάζομαι γνωρίζετε το άρθρο και γνωρίζετε τι έγινε αφού ήσασταν ε, παρόν και οπότε φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι έγινε. Τώρα έχουμε τα πρακτικά της κοινής συνεδρίασης, επίσης έχουμε και τα κείμενα τα οποία εγκρίθηκαν. Έχετε κάποια ένσταση, κάποια παρατήρηση, ιδάλλως εγκρίνονται τα πρακτικά. Έχουμε τώρα μία έγγραφη δήλωση υπαριθμών 8 20, για το 2015 όσον αφορά το ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, προσπάθειά μας ε, για την καταπολέμηση της πολιομυρίτητας τρέχουμε έχουμε κυρία Μακάβαν, η οποία επίσης έχει αναλάβει να συγκεντρώσει κάποιες